Τώρα ερχόμαστε στις ψηφοφορίες και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα έχουμε απλοποιημένη διαδικασία για την έκθεση του κυρίου Hans Peter Marking ονομαστική αξία για τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ και πρόκειται για να κυκλοφορήσουν. Ονομαστική ψηφοφορία ξεκίνησε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Τότε λίγη ψηφοφορία. ενεκρίθη. Σύμφωνα με ε, την ημερήσια διάταξη έχουμε απλοποιημένη διαδικασία και για την έκθεση Μπορσελίνο για τη στρατηγική εξωτερική ασφαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινά ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τώρα έχουμε επίσης μαπροποιημένη διαδικασία την έκθεση De Jong, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Ξεκινά η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Λίγη ψηφοφορία. Ενεκρίθη. Επίσης με απροποιημένη διαδικασία θα ψηφίσουμε την έκθεση Ριγκογέν Περές για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευαλώτων καταναλωτών. Ψηφίστε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Πέτερ Μάρτιν για την έκδοση κερμάτων των ευρώ. Εξετάζουμε την πρόταση κανονισμού. Έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ποιος μπορεί να τις δεχθεί ο ε, μπλοκ. Ε, υπέρ κατά ενεκρίθησαν και τελειώσαμε με το δεύτερο μπλοκ και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινά τώρα. Ψηφίσατε. Λίγοι. ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία. Ακολουθεί η έκθεση Μπουσουτήλη για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Εξετάζουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Υπάρχει μία τροπολογία για την παράγραφο 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. Θέλει κάποιος να υπάρξει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινά. Λίγη. Ε, παρακαλώ για ξαναψηφίστε διότι υπήρξε ένα πρόβλημα τεχνικό. Παρακαλώ να ψηφίστε και πάλι δεύτερη φορά. Ψηφίσατε. Έληξε. η τροπολογία ε, νεκρήθη. Και τώρα ερχόμαστε στο σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγοι. Ενεκρίθη. Ερχόμαστε στην έκθεση Μποσκούρτ για την προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020. Ε, υπάρχει, ε, θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα, η τροπολογία 9 περίφθη και ψηφίζουμε συνολικά 7 τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα ψηφίσουμε την παράγραφο 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 7. Υπέρ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι την τροπολογία 7. Λίγη. Ενεκρίθη η τροπολογία. Ερχόμαστε τώρα στην παράγραφο 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. Παράγραφο 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά ενεκρίθη 49 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 52 και πάλι σε δύο τμήματα ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης παράγραφος 57 ονομαστική ψηφοφορία ξεκινά τώρα ψηφίσατε όλοι λίγοι ενεκρίθη. Παράγραφος 61 και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. ενεκρίθη το ψήφισμα και τώρα ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκίνησε. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ενεκρίθη. Τώρα ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Γκουρμάη σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ψηφίζουμε ε, για την... Ε, ε, για την έκθεση αυτή η κυρία Γκουρμάη έχει το λόγο Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει από τις πρώτες, ισχύει από τις 1 Απριλίου, πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ε, τις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη πρωτοβουλία οργανώθηκε στις 9 Μαΐου στην ημέρα της Ευρώπης και βλέπω ότι πολλοί πολλοί από εσά έχουν δείξει τόσο ενδιαφέρον για αυτή την πρωτοβουλία και παρακαλώ να θεωρηθούν οι ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν επίκεντρο της εκθέσεώς μου για να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρξουν ορισμένα τεχνικά σημεία και θα ήθελα να προχωρήσουμε ε, και ε, να ε, υπάρξει, ε, υπάρξει θετική στήριξη της τροπολογίας 4 και αρνητική της 5. Επίσης προτείνω τα εξής. Εάν ισχύσει η τροπολογία ε, θα υπερψηφίσω το τρίτο μέρος της τροπολογίας 1 και 3 αλλά εάν η τροπολογία 5 ισχύσει χωρίς το 3 τότε θα προχωρήσουμε ελπίζω ότι με παρακολουθήσετε και θα επανέλθω όταν θα υπάρξει ηλεκτρονική ψηφοφορία ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη θα δούμε αν εγώ μπόρεσα να σας παρακολουθήσω λέει ο πρόεδρος ε, προχωρούμε στην τροπολογία 5 5.1. Έχουμε έξι τμήματα. Πουθενά δεν προβλέπεται ονομαστική ψηφοφορία, οπότε καταρχήν ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται η κυρία Γκορμάη έχει το λόγο θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ Ευχαρίστως να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για το τμήμα 2. Ξεκινά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία. Ερχόμαστε στο τρίτο τμήμα της τροπολογίας 5. Κυρία Γκορμάη. Λυπάμαι πάρα πολύ είχα ζητήσει ε, και ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία για το 3 αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το επόμενο. Το πέμπτο δηλαδή. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το τρίτο ο, τμήμα της τροπολογίας 5. Ξεκινά ηλεκτρονική επαλήθευση και και Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ενεκρίθη. Ερχόμαστε στο τέταρτο τμήμα της τροπολογίας 5. Ποιος είναι υπέρ, διανατάσσεως χειρός. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Ενεκρίθη. Ερχόμαστε στο πέμπτο τμήμα το οποίο να πεσύρθει. και ερχόμαστε στο έκτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινά ψηφίσατε όλοι έληξη ψηφοφορία υπερψηφίστηκε Τώρα μου λέγεται ότι πρέπει να ψηφίσουμε το πέμπτο τμήμα της τροπολογίας 1, αυτό που είχε αποσυρθεί από το ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του πέμπτου τμήματος της τροπολογίας 1 της Επιτροπής. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τώρα Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 των φιλελευθέρων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. 2. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, επίσης ενεκρίθη. Ερχόμαστε σε ονομαστική ψηφοφορία όλου του, όλης της εκθέσεως. Ποιος ε, ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. με μεγάλη πλειοψηφία ενεκρίθη και συγχαίρω την κυρία Γκουρμάρη. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Έχουμε τώρα βέβαια τις επεξηγήσεις ψήφου.